στην ημερήσια διάταξη όπως εγκρίστηκε από τη συνδιάσκεψη των Προέδρων 4 Μαρτίου. Ερχόμαστε λοιπόν στο 137. Τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν υπάρχουν μεταβολές στην ημερήσια διάταξη, στο σχέδιο αυτό δηλαδή. Όσον αφορά όμως την Τετάρτη, για να πάμε στην Τετάρτη. κυρία Ρεμπέκα Χάιμς, θα υποβάλει ένα ψήφισμα εκ μέρους των Πρασίνων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ζητήσαμε για άλλη μια φορά το θέμα της έγκρισης ε, της ε, γενικά τροποποιημένης πατάτας φλόρα να τεθεί για άλλη μια φορά στη Μέση διάταξη για τους εξής λόγους. Τώρα που στην Κομισιόν επίτροπος που είναι αρμόδιος για τους τρογενικά τροπημένους ε, οργανισμούς είναι ο επίτροπος αρμόδιος για ε, την υγεία ε, θεωρούν οι πολίτες ότι υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή στην έγκριση αυτών των τροπι... γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Τον ήθετο όμως συμβαίνει και μου φαίνεται πραγματικά σκανδαλώδες ότι ο Επίτροπος, ο υπεύθυνο για την Υγεία, α, έχει παραβλέψει όλες τις επιφυλάξεις του Διεθνούς, της διεθνούς Οργάνωσης Υγείας για τη Ματάτη. Και θα να σας πω, στην τελευταία θητεία μεταξύ Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής υπήρχε έντονη διαφωνία όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης, γιατί πολλά κράτη-μέλη δεν συμφωνούσαν με <clears throat> τις προσπάθειες έγκρισης που είχαν προωθήσει ιδίως ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Μπαρόζο και είχε συμφωνηθεί να υπάρξει μια νέα πιο ε, περιστατωμένη διαδικασία έγκρισης. Πού είναι αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι εμεί στην πλειοψηφία των πολιτών είμαστε κατά της έγκρισης αυτής της πατάτας και θα πρέπει νομίζω να γίνει αυτή η συζήτηση για την έγκριση αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας κύριε Πρόεδρε. Ε, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για την ψηφοφορία να γίνει ονομαστική κλίση. Πρόεδρος, θα ήθελε κάποιο να ταχθεί υπέρ αυτή τη πρόταση, Ο κύριο Σούλτ. Είσαστε κατά, καλά. Μετά λοιπόν εσείς. Ποιος θα υποστηρίξει την πρόταση πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πέρα από τις αξιολογήσεις των ε, μεμονωμένων βουλευτών ή των πολιτικών ομάδων, θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο σε ένα τόσο σημαντικό θέμα να αποφανθούμε. Διότι συζητάμε τόσα πράγματα τα οποία είναι πολύ μακρινά από εμάς, ενώ αυτό το θέμα αφορά άμεσα εμάς, το εκλογικό μας σώμα και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ κατά ο κύριος Σούλτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, εγώ συμμερίζομαι τις επιφυλάξεις της συναδέλφου Χάμς και σε πολλά κράτη-μέλη βλέπουμε πολύ αντιφατική συζήτηση του θέματος. Γι' αυτό ήδη στη διάσκεψη των Προέδρων την περασμένη εβδομάδα είχα πει αυτό που θέλω να επαναλάβω εδώ και τώρα. Νομίζω ότι δεν θα μας οδηγήσει πουθενά να κάνουμε τώρα στα γλίγορα μια συζήτηση χωρί ψηφισμά που θα εξαφανιστεί. Θα πρέπει να αναθέσουμε στην αρμόδια επιτροπή να ορίσει έναν εισηγητή που θα ασχοληθεί με όλη τη διαδικασία και με την τεχνολογία της διαδικασίας έγκρισης. Η έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής ε, έγινε μετά από 8 χρόνια μελέτης και βάση σε ευρωπαϊκό δίκαιο και η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία όπως προβλέπετε. Ε, θα πρέπει να ρωτούμε κατά πόσον αποφάσεις τέτοιου εύρους δεν θα πρέπει να υποβάλλονται στην απόφαση του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό θα ήταν καλό να ορίσουμε εισηγητή που θα εξετάσει τον μηχανισμό και ενδεχομένως να υποβάλει μία έκθεση και να πετύχει νομοθετική πλειοψηφία εδώ που θα υποχρεώσει την Εκτελεστική Επιτροπή. Κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, δύο δευτερόλεπτα υπομονή σας παρακαλώ. Καθένα εδώ λέει ό,τι θέλει, γιατί να μην μιλήσω. Λοιπόν, λέω, να έχουμε το στόχο να πείσουμε να υποχρεώσουμε μάλλον την Κομισιόν μέσα σε ένα χρόνο να μας υποβάλει μια νομοθετική πρόταση. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο από μια γλίγορη συζήτηση αυτή τη στιγμή εδώ και τώρα. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Σούλτς. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ να θυμόσαστε ότι μπορείτε να πάρετε το λόγο για ένα λεπτό για να ταχθείτε υπέρ ή κατά της πρότασης. Λοιπόν, σας παρακαλώ, σεβαστείτε το χρόνο αυτό, να είστε πειθαρχημένοι, να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό. Ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε την πρόταση της ΓΚΟΕ και των Πρασίνων για ονομαστική ψηφοφορία. Το αίτημα αυτό πρέπει τώρα να ψηφιστεί. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης της ε, κυρίας Ρεμπέκα Χάιμς. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ονομαστική είναι, είπαμε, οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. ...82 υπέρ, 182 κατά, 15 αποχές. Συνεπώς η πρόταση απορρίπτεται. Συνεπώς, η ημερήσια διάταξη για την Τετάρτη παραμένει ω είχε. Δεν υπάρχουν μεταβολές για την Πέμπτη και συνεπώς η ε, ημερήσια διάταξη ολη τη εβδομάδας εγκρίθηκε. Το επόμενο θέμα μας είναι η δήλωση του Προέδρου σε σχέση με την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα είναι διαφορετική από την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας που θυμόμαστε τουλάχιστον στις κεντρικές και ανατολικές χώρες της Ευρώπης. Δεν δίνουμε μόνο λουλούδια πια στις κυρίες. Ε, συζητείται συνεχώς η ισότητα των φύλων, η υποστήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το Ευρωκοινοβούλιο θέλει και αυτό να συμμετάσχει σε αυτή την έντονη συζήτηση στα καυτά θέματα αυτά. Η Επιτροπή λοιπόν των Δικαιωμάτων της Γυναίκας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Το 2009 τον Νοέμβριο υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα κάνοντας έκκληση προς τα κράτη-μέλη να ενεργήσουν κατά της βίας κατά των γυναικών. Θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί του υπολείπου κόσμου σε αυτόν τον τομέα. Σήμερα οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη διότι ε, ξέρουμε ποιες είναι οι δημογραφικές τάσεις μεν στην Ευρώπη, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποβαίνει σε βάρος των γυναικών. Οι γυναίκες πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται και να μπορούν να συνδυάσουν τον οικογενειακό βίο με τη σταδιαδρομία τους. Συνεπώς πρέπει να ε, τους δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν ε, νηπιαγωγεία για να φροντίζουν τα παιδιά τους και οι γυναίκες που θέλουν να μείνουν στο σπίτι τους θα πρέπει να μπορούν να το πράξουν αυτό μέσω ενός σωστού συστήματος φορολόγησης. Δηλαδή, ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ισότητα σε όλα τα θέματα. Οι διακρίσεις στην κοινωνία, στην σταδιοδρομία πρέπει να ανήκει πια στο παρελθόν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι άντρες και οι γυναίκες είναι ίσοι από κάθε πλευρά και το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει και αυτό να συμμετάσχει σε αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες θα ήθελα οι γυναίκες στο Ευρωκοινοβούλιο να μην αισθάνονται ότι είναι υποκείμενα διακρίσεων. Ελπίζω λοιπόν ότι στο Ευρωκοινοβούλιο θα αποκτήσουμε όλο και περισσότερο, περισσότερες βουλευτίνες. Τώρα, θα μιλήσουν οι πολιτικές ομάδες το, από το ΕΛΚ, η κυρία Βότονσκολ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε σήμερα, είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Εκατοστή επέτειος μάλιστα είναι. Ε, μέρα γιορτής έχουμε πετύχει πολλά πράγματα.